Συνεχίζουμε τώρα με την τελευταία έκθεση στην ημερήσια διάταξη του κυρίου Γκρασαμόρα για την πολυγλωσία. Ένα κοινό εγχείρημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο «Πολυγλωσία, ένα θετικό στοιχείο για την Ευρώπη και μια κοινή δέσμευση» έχει οδηγήσει σε μια πληθώρα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Κομισιόν, την Επιτροπή Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου θίγεται το θέμα τη πολυγλωσία από πολλέ οπτικέ γωνίε. Η δική μου έκθεση υπενθυμίζει τι θέσει που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποστηρίζει την θέση τη Κομισιόν ότι είναι ένα πραγματικό πολιτιστικό <clears throat> και κτημένο και ένα ε, ατού στον ανταγωνισμό η πολυγλωσία. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης πολυγνωσίας και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γλώσσα είναι παράγον κοινωνικής ενσωμάτωσης, είναι παράγον διαλόγου με άλλες χώρες του κόσμου, ιδίω με τις χώρες με τις οποίες έχουμε κοινή γλώσσα για ιστορικούς λόγους οι ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να υποστηριχθεί η μετάφραση στο τεχνικό και στο ε, λογοτεχνικό επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε πολυγλωσία στα πολυμέσα, να έχουμε ανάπτυξη της ε, γνώσης όλων των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης άλλων γλωσσών οι οποίες ομιλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι κλασικές γλώσσες, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Η γνώση των γλωσσών είναι σημαντική, αλλά η βάση όλων αυτών είναι η γνώση της μητρική γλώσσας. Θα πρέπει οι γονείς των παιδιών να μπορούν να διαλέξουν τη γλώσσα στην οποία θα εκπαιδεύονται τα παιδιά τους σε χώρες όπου υπάρχει παραπάνω από μία επίσημη γλώσσα ή όταν συνεπάρχουν μία επίσημη γλώσσα και περιφερειακές γλώσσες. Δεν μπορεί κανείς να αποστελθεί του δικαιώματος παιδεία στη μετρική του γλώσσα. Θέλω να τονίσω επίση στην έκθεσή μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε και τη σημασία των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θυγούν αυτές οι γλώσσες και δεν είναι η υποστήριξη πολυγνωσίας ασύμβατη με αυτές. Εδώ υπάρχει επίσης και μια πρόταση των φιλελευθέρων, των σοσιαλιστών και των πρασίνων που ακυρώνει αυτά τα τρία σημεία τα οποία προανέφερα. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που θα πρέπει να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ περιλαμβάνονται τα δικαιώματα γλωσσών όπως η καταλανική, η βασική και άλλες που έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ελπαίς έχει μια ειδική ε, σελίδα που αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η παροχή εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια αναλλακτική λύση σε όλα αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός των εθνικισμών και είναι επίση απαράδεκτο να υπάρχει η παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και να θίγεται η αρχή της ε, επικουρικότητας. Πρέπει επίσης η θέση μας να βασιστεί στα προηγούμενα κειμένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να επιθυμίσω σε όλους ότι η εναλλακτική αυτή λύση, η πρόταση των φιλελευθέρων σοσιαστών και πρασίνων, θα πρέπει <clears throat> να ε, απορριφθεί και να υποστηρίξουμε υπέρ της πρότασης Επιτροπή Πολιτισμού που έγινε δεκτή σχεδόν με ομοφωνία μοναχά τρει ψήφου κατά και δύο εποχέ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υποστηρίξουμε τη σημασία τη δημοκρατία και του πλουραλισμού, να μην υπάρξει αποκλεισμό δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Μισελ, έχετε το λόγο και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάσα Μούρα για την έκθεση αυτή κατά πρωτοβουλία σχετικά με την πολυγλωσία. Η έκθεση αυτή στηρίζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τονίζει την σημασία της προωθήσεως των γλωσσών για να καλύψει όλες τις πτυχές της κοινωνίας ε, μέσω της γλωσσικής διάστασης και να βοηθήσει την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των ατόμων και ε, την πρόθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των στενότερων σχέσεων με τρίτες χώρες. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η πολυγλωσία επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών δεδομένως της ε, συνεχούς μετακινήσεως και της προωθήσεως της ε, παγκοσμιοποίησης. Η ε, προώθηση της γλωσσικής γλώσσας συν δύο παραμένει το επίκεντρο της πολυγλωσσίας και η μέθοδός μας βασίζεται σε, αυτή, αυτό το και εκτιμένο κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και ε, τα ευάλωτα άτομα της κοινωνίας που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδέ τους και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ε, γνώσεις ε, όλων των ηλικιών. Χαίρομαι που προσφέρεται αυτή η δυνατότητα και πιστεύω ότι η παιδεία είναι πολύ βασική. Η νέα τεχνολογία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τα άτομα και τις ομάδες αυτές που έχουν ειδικέ ιδιομορφίες και η διαβίου μάθηση στην Ευρώπη καλύπτει όλες τις γλώσσες και τις περιφερειακές και ε, τις μικρότερες γλώσσες που μιλούνται σε άλλα σημεία του κόσμου. Κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε τις γλωσσικές ανάγκες των ε, πολιτών μας και με την ε, μετανάστευση είναι βασικό να προωθήσουμε τις εθνικές γλώσσες για να μπορεί κανείς να ενταχθεί στην κοινωνία αλλά θέλω να σας πω ότι τα κρατη μερη είναι αυτά τα οποία λαμβάνουν απόφαση σχετικά με τις ε, γλωσσικές πολιτικές ακόμη και για τις περιφερειακές ή τις μειονεκτικές ε, γλώσσες και χαιρετίζω την προσέγγιση του Ευρωκοινοβουλίου στην πολυγλωσσία. Ευχαριστώ. Και σε αυτή την, έκθεση, αυτή την έκθεση θα την ψηφίσουμε αύριο. Εξαντλήσαμε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο 3η 24 Μαρτίου από τις 9 η ώρα το πρωί σε τρεις συνεδρίες και ε, λίγη συνεδρίαση. Καληνύχτα σε όλους.